και ε, κύριο Τζανόνι από πλευράς Φιλελευθέρων. Ευχαριστώ όλους σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Συγχαρητήρια η γραπτή δήλωση 0037-2011 που έχουν υποβληθεί από τον κύριο Δανέλη και λοιπόν όσον αφορά το σύμφωνο των νήσων έχει δεχτεί τις ε, υπογραφές ε, της πλειοψηφίας των μελών που συνθέτουν το Κοινοβούλιο και επομένως σύμφωνα με το άρθρο 123 ε, θα προωθηθεί δεόντως και επομένως θα αναφερθεί στα υιοθετημένα εγκριμένα κείμενα. Ο κύριος Δανέλης παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι αισιόδοξο αγαπητοί συνάδελφοι να εκφράζεται τη κοινή μας βούληση για ενίσχυση της συνοχής, η έμπρακτη στήριξη στην ισιωτικότητα, καθώς επίσης και η προώθηση της βιώσιμης περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά ανάπτυξης. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους καλούς συναδέλφους ε, καρβάλιο ουτζίας μαυρονικόλα σμιθ και όλους εσάς που συνυπογράψατε την δήλωσή μας καθώς επίσης τους συνεργάτες μας και την Ίνγκε και τον αλεσάνδρο. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια και σε εσά κύριε Δανέλη και επομένως τώρα θα ξεκινήσουμε με τις ψηφοφορίες. Έκθεση Λουί Μισελα σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό ε, για θέσπιση